Ladies Κυρίες και κύριοι. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ξεκινήσει η πρώτη ψηφοφορία σε 10 δευτερόλεπτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω δύο ανακοινώσεις να κάνω πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Η πρώτη είναι η εξής. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, επαναλαμβάνω. Η πρώτη ανακοίνωση είναι η εξής. Ο πρόεδρος έχει λάβει από την ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών αίτημα αλλαγής ε, ονόματος σε επιτροπή και σε αντιπροσωπεία. Οι αλλαγές θα υπάρχουν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και αν δεν έχετε παρατηρήσεις να υποβάλλετε πριν την έγκριση των πρακτικών οι αλλαγές αυτές θα θεωρηθούν εγκριθήσεις. Η δεύτερη ανακοίνωση είναι η εξής. Σύμφωνα με το κανόνα 152 εδάφιο 2 και σύμφωνα με ναι. και σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες σας προτείνω την εξής αλλαγή στην ημερήσια διάταξη